και έχουμε τώρα ένα αποτελεσματικό νομοθετικό μέσο εφόσον το ψηφίσει το Κοινοβούλιο την Τετάρτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περαιούται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει Τετάρτη 12. Προχωράμε με κάποιες ανακοινώσει Πρώτον, έλαβα από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές Έτηση ανάκληση τη ασυλία του, κυρίου, του βουλευτού κυρίου Έλμαρ Μπρόκ μετά από αίτημα τη αγγελία του Μπίλεφελτ. Βάσει του άρθρου 6 παραγωγή 2 του κανονισμού το αίτημα ε, παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, την νομική επιτροπή. Επίση, η Προεδρία έλαβε από την ομάδα τη Προεδρική Συμμαχία σοσιαλιστών και δημοκρατών στο Κοινοβούλιο από την ομάδα των φιλελεύθερων και από την γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών αιτήματα ορισμού βουλευτών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και αντιπροσωπείε. ο κατάλογος των ε, υποψηφιωτήτων θα υποβληθεί στα πρακτικά της παρούσης ε, ε, ημερήσια της των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης και θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει. Προχωρούμε τώρα. Παρεμβάσεις ενός λεπτού για θέματα πολιτικής σημασίας. Παρακαλώ να τηρήσετε με απόλυτη το σεβασμό το ένα λεπτό. Ο κύριος Νίκουλαεσκου, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της προσχώρησης της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Θεωρώ ότι δεν πρέπει ε, να ε, αναμειγνύουμε τα θέματα μεταρρύθμισης δικαιοσύνης με τα θέματα του χώρου Σέγγεν. Η Ρουμανία είναι έτοιμη και πληρεί τις τεχνικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να αποτελούν και το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση. Η Ρουμανία δεν είναι χώρα, ούτε θα είναι χώρα εξαγωγής εγκληματιών και δεν μπορούμε να δεχθούμε το να στιγματίζεται ε, η Ρουμανία στο εξωτερικό και ε, ο λαός της Ρουμανίας. Η ψηφοφορία την επόμενη άνοιξη πρέπει να είναι πολιτική ψηφοφορία που θα βασίζεται σε αντικειμενική αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόπα έχει το, λόγο. Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφή στη Λισαβόνα γενιάζει μια νέα εποχή στην προσπάθεια τη συμμαχία να αντιπεξέλθει στι νέε προκλήσει σημαντική είναι στο πλαίσιο αυτό η αναγνώριση της μοναδικότητας της εταιρικής σχέσης συμμαχίας με την ευρωπαϊκή ένωση όπως και της ανάγκης για συνεχίσεις σε όλες τις πτυχές ευρωπαϊκής ασφάλειας. σε κάθε περίπτωση η συνεργασία των δύο οργανισμών πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια συμπληρωματικότητα αλλά και σεβασμό στην αυτονομία του καθενός εκ των δύο ιδιαίτερη σημασία έχει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με συνέργειες και να αποφύγουμε αλληλοεπικαλύψεις κυρίως σε θέματα πολιτικών αποστολών που θα αποτελούσαν μια μεγάλη σπατάλη προσωπικού και ενέργειας για τα κράτη μέλη τόσο της ένωσης όσο και του νατο και αυτό είναι κομβικό για την αποτελεσματικότητα αλλά και την εξοικονόμηση πόρων ο τρόπος με τον οποίο θα κατοχυρωθεί η θεσμική συνεργασία των δύο οργανισμών η δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού διαβούλευση, που έγκαιρα θα προσδιορίζει τον τρόπο και τα μέσα κοινή δράση είναι πολύ σημαντικός. θα ήθελα να ζητήσω να γίνει μια σε βάθο συζήτηση για το θέμα αυτό. ευχαριστώ. Στις 28 Νοεμβρίου στην Μολδαβία θα γίνουν πρώτες εκλογές, διότι η Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι στην κυβέρνηση ένα χρόνο και, και έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία πέδειξε τη βούλησή της να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Οδό η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα δεδομένα υποστηρίζει οικονομικά και πολιτικά την Μολδαβία. Ελπίζω ότι οι κυριακάτικες εκλογές θα ξεκαθαρίσουν απόλυτα το δρόμο της Μολδαβίας ως μια πλήρη δημοκρατία, ένα κράτος δικαίου και η λειτουργική οικονομία της αγοράς και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάποτε ελπίζω να γίνει μέλος. Και η Μολδαβία ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έχει το λόγο. Θέλω να καταγγείλω μια θλιβερή συμπεριφορά της Γραμματείας της Επιτροπής Περιφερειών σε σχέση με μια έκθεση φωτογραφίας που οργανώνει ο εκτοπισμένος Δήμος της Κερίνιας της κατεχόμενης σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα πόλης στην δική μου την πατρίδα την Κύπρο. Στις φωτογραφίες που εκτίθενται απεικονίζεται ανάγλυφα η καταστροφή εκκλησιαστικών και άλλων μνημείων της τρισχιλιετούς ιστορίας της Κερίνιας ο στόχος των καταστροφών έκδηλος να αφανιστεί οτιδήποτε που μαρτυρεί ότι αυτή την πόλη την κατοικούσαν άνθρωποι με ελληνικό πολιτισμό και χριστιανική πίστη άνθρωποι που εκδιώχθηκαν από τι αιστείε του με τη βία που κατορθώνουν και ξεριζωμένοι στην προσφυγιά να απλώνουν μετά από 36 χρόνια τι ρίζε του στην κερίνια. αυτή την έκθεση θα την άνοιγε ο Γενικό Γραμματέα τη Επιτροπή περιφερειών ο οποίος τελικά δεν εμφανίστηκε υποκύπτοντας τις πιέσεις της κατοχικής δύναμης της τουρκίας γιατί η έκθεση αναφέρεται στην εισβολή της χώρας αυτής στην κύπρο το 1974 και την καταστροφή της πολιτιστικής της κληρονομιάς από τους εισβολείς. μάλιστα απαιτήθηκε από τη γραμματεία της επιτροπής το ξύλωμα της έκθεσης αυτής. καταγγέλλω αυτή την απαράδεκτη ενέργεια. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διάσωση της Ιρλανδίας μάλλον δεν θα είναι η τελευταία που θα συμβεί στην Ευρωζώνη παρότι όλοι αυτό ισχυρίζονται. Παρά την χρήση του, χρέου, του χρέους το, όλοι επιμένουν να πούν ότι το πρόβλημα της Ιρλανδίας είναι διαφορετικό από ό,τι πριν από 7 μήνες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν οφειλόταν στη, στην δημοσιονομική ανευθυνότητα και στη διαφθορά, ενώ στην Ιρλανδία ε, οφείλεται στην ε, συμπεριφορά των τραπεζών. Η Πορτογαλία προσπαθεί να μην πνιγεί όπως και η Ισπανία τι είναι το κοινό στοιχείο αυτών των χωρών, ότι το ενιαίο νόμισμα, τους δεν, το νόμισμα δεν τους ταιριάζει. Ε, όλα τα έχουμε ρίξει σε ένα καλάθι και το πρόβλημα που υπάρχει είναι σαφές. Οι χώρες που έχουν ε, το δικό τους νόμισμα, οι οποίες μπορούν να ελέγξουν το νόμισμά τους και να κάνουν ε, συναλλαγές με τους εταίρους τους, είναι σε καλύτερη θέση υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθεί το συνολικό κεφάλαιο της ε, Ευρωπαϊκής ε, ε, της Ευρωζώνης και καλά είναι να περάσουμε σε ευθανασία. Ο, ο κύριος Χέρεν Χάουζερ. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε και η Ιρλανδία ε, ένα τομέα που πρέπει να φροντίσουμε και μας ενδιαφέρει η δημιουργία χρήματος. Η δημιουργία χρήματος από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες ε, τροφοδοτούνται μεγάλες ποσότητες χρήματος στο σύστημα δημιουργώντας ε, πληθωρισμό και δημιουργώντας και μαζικά χρέη. Έχουμε μια συστημική κρίση την οποία δεν μπορούμε να λύσουμε επενδύοντας δισεκατομμύρια σε ένα ε, ήδη άρρωστο τραπεζικό σύστημα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια μεταρρύθμιση του συστήματο δημιουργία χρήματο. Το σύστημα δημιουργία χρήματο θα πρέπει να το αναλάβει ο δημόσιο τομέα. μέσω των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της δημιουργίας χρήματος να έχουμε κάτι συμβατό με την οικονομία της αγοράς. Βέβαια, ε, για τόσο ε, ριζικές αποφάσεις ε, ε, χρειάζονται ριζικές αποφάσεις ε, που θα αφορούν και τον τραπεζικό τομέα και μπορούν να βοηθήσουν και το Κοινοβούλιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Τόκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά για την 95η επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους. Με απόφαση που λήφθηκε και σε συνέχεια της απόφασης αυτής το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρήσει να θυμηθεί ότι 1,5 με 2 εκατομμύρια Αρμενίων σφάχτηκαν και θανατώθηκαν μια κατάσταση αντίστοιχη με το ολοκαύτωμα ή τις δολοφονίες στην Σοβιετική Ένωση όπως και με τις φαγές ε, άλλων χριστιανικών πληθυσμών από τις Οθωμανικές αρχές. Πολλές χώρες ήδη έχουν αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν πέρασε ένα τέτοιο θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο Μπούζεκ να υπάρξει αναγνώριση της ερμενικής γενοκτονίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρηθεί ως γενοκτονία και να αποτελέσει η αναγνώριση υποχρεωτική δέσμευση της γενοκτονίας, ε, ε, υποχρεωτική δέσμευση της Τουρκίας. Ο κύριος Μπλουμ έχει το λόγο. Κύριε Μπλουμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα άτομα από 18-27 ετών στη Ρουμανία θεωρούν ότι έχει επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση και μόνο 33% των νέων στη Ρουμανία λένε ότι δεν θέλουν να μεταναστεύσουν. Με την πολιτική περικοπών των μισθών η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι ότι επιταχύνει τη διαρροή εγκεφάλων. Υπάρχουν νέοι που έκαναν τις σπουδές τους στο εξωτερικό και είτε φεύγουν είτε δεν βρίσκουν απασχόληση. Ακόμη και αν έχουν την απαραίτητη εμπειρία και την ε, βούληση να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ε, οικονομίας της Ρουμανίας. Ε, η κυβέρνηση στο Βουκουρέστι πρέπει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και οι υπότροφοι της Ρουμανίας ε, ε, που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν όλοι μας την υποστήριξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αλληλευτικά σκάφη που αλλιεύουν στον Ινδικό υφίστανται ένα κύμα πειρατικών επιθέσεων. Δέκα επιθέσεις την, την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Ροσμπακάν, του Ροσάτε, στην, στην ακτή του Ινδικού γενικότερα και όλο και μακρύτερα από την ακτή, διότι οι πειρατές χρησιμοποιούν όλο ένα και μεγαλύτερα ε, σκάφη. Ε, πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός διότι ο Ναφός σε καμία από τις επιθέσεις δεν ε, επιτέθηκε και δεν ξέρουμε πώς να απαντήσουν στις ε, προειδοποιήσεις αυτές. Θα πρέπει να υλοποιηθεί το ψήφισμα που υιοθετήσαμε την περασμένη, τον περασμένο χρόνο στο Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παρέμβαση των, ε, των και της Ένωσης μέσω της Αταλάντης αλλά και μεγαλύτερη εμπλοκή των παράκτιων χωρών. Η πειρατεία έχει συνέπειε στα λευτικά σκάφη, στην αλευτική δραστηριότητα. Οι χώρε με τι οποίε ε, έχουμε ε, συμφωνίες ε, αλευτική συνεργασία πρέπει επίσης να μετάσχουν στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ρώση έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταγγείλω στο Κοινοβούλιο αυτό που έγινε με την έκθεση για την προώθηση ε, στην, ε, της κατεχόμενης Κύπρου στην Επιτροπή Περιφερειομίας έκθεσης από τις 27 έως 29 Νοεμβρίου. Στις 17-19 ε, Νοεμβρίου, στις 17 Νοεμβρίου μετά την, το ξεκίνημα ο, ο εκπρόσωπος της γραμματείας ζήτησε να κατέβει η έκθεση λέγοντας ότι οι πίνακες έδειχναν διαφορετικ, περίχαν διαφορετικές λεζάντες από αυτές που είχαν συμφωνηθεί ζητήθη, εγώ ε, έλεγξα και διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ της άδειας που είχε δώσει και των εκθέσεων. Επιπλέον, ο υπεύθυνο τη έκδοση ε, πήρε εντολή να διαγράψει τη λέξη κατοχή και εισβολή. Μίλησα με τον επικεφαλής για να μάθω τι έγινε, αλλά ούτε ο υπεύθυνο ούτε οι συνεργάτες του δέχτηκαν να μιλήσουν μαζί μου. Λίγες ώρες μετά την καταγγελία των γεγονότων αυτών, ξανά άνοιξε η έκθεση. Συνάδελφοι, αυτό που συνέβη στην Επιτροπή Περιφερειών είναι πολύ σοβαρό γεγονός βλαπτικό ενός κράτους μέλους της Ένωσης. Ο κύριος Βάντιμ Τούντορ. Ευχαριστώ. a Europei. A fost rău cu dictatura comunistă, e η Ρουμανία έχει γίνει το άγριο σύνορο της Ευρώπης. Ήταν δύσκολο κατά τη διάρκεια της ε, ε, Σοβιετικής δικτατορίας, αλλά τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. 5.000 δολοφονίες των οποίων ε, οι υπεύθυνοι δεν έχουν συλληφθεί έγιναν από τον Ιανουάριο του 1990 μέχρι τώρα ε, στη Ρουμανία. Είναι παράδεισος ε, των μαφιόζικων οργανώσεων αλλά επίσης είναι και χώρος διακίνησης, χώρο ελευθερίας για παιδεραστές και μια σειρά από άλλους κακοποιούς. Το Δεκέμβρη του 1990 1990 ε, ε, ε, υπήρχε ο τουρισμός για το Δράκουλα και τώρα δεν ξέρουμε πώς να τον ξεφορτωθούμε. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το τελευταίο καιρό ένα μαύρο σύννεφο όλο και πυκνότερο απλώνεται στην Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε. Η εκλογική άνοδος σχηματισμών και κομμάτων μιας μυσαλόδοξης, ξενοφοβικής και πολύ συχνά ρατσιστικής άκρας δεξιάς έχει σημαδέψει τι πολιτικέ εξελίξει σε πολλά κράτη μέλη ακόμα και στη σουηδία. είναι ιονό που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το διωγγούμενο μεταναστευτικό πρόβλημα συνενώνονται σε ένα δηλητηριώδε μείγμα που τρέφει άκρα και ακρότητε. πρόκειται αναμφισβήτητα για εξαιρετικά πολύπλοκο και δυσεπίλητο πρόβλημα. γι' αυτό τα κεντρικά πολιτικά κόμματα τη ευρωπαϊκή κέντρο δεξιά και σοσιαλδημοκρατίας και εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα και οι σοσιαλιστές έχουν μια σοβαρή ευθύνη και αποστολή να διώξουν το σύννεφο πριν αυτό φέρει καταιγίδα. οφείλουν να εξαντλήσουν τις δυνατότητες συνεννόησης και συντονισμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως το μεταναστευτικό τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες του καθενός χωριστά. εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οφείλουμε κυρία πρόεδρε να αναλάβουμε μια νέα ισχυρή κοινή πρωτοβουλία κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην ευρώπη της κρίσης. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο δεν ξέρω αν τα μάτια της Ευρώπης είναι στραμμένα στην οικονομική κρίση της χώρας μου, η οποία κρίση προκλήθηκε από την πλεονεξία, την καθαρή πλεονεξία όλων των οικονομικών παραγόντων, οι οποίοι πρέπει να, τε, θεωρούν υπεύθυνοι. Βεβαίως όμως η έλλειψη ρύθμισης του τραπεζικού τομέα προκάλεσε και αυτή την κρίση. Αυτό ισχύει στην Ευρώπη. Η Κομισιόν ε, απείλαξε τις, τις τράπεζες ε, Πώς συνέβη αυτό. Είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος, εξαιρετικά εξοργισμένος που έφτασε στο σημείο αυτό η χώρα μου. Ποια είναι η αλληλεγγύη που δείχνουν οι συνάδελφοι σε όλη την Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδία είναι ένα κυρίαρχο κράτος και οποιασδήποτε επιταγές από την Ευρώπη για την φορολογική πολιτική της Ιρλανδίας θα είναι επικίνδυνε όσον αφορά την μεταχείριση των μικρότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άρκιν. Κύριε Χάρκιν, θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για την τρέχουσα οικονομική κρίση από διαφορετική ε, όμω οπτική γωνία. Ακούσαμε τον κύριο Τρισέ και τον Όλυ Ρεν να μιλούν ε, για την οικονομική ανευθυνότητα και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία ε, και το, την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αν ακούσουμε τα ευρήματα από τη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου που σήμερα δημοσιεύθηκε, η μελέτη αυτή ζήτησε τη γνώμη πάνω από 27.000 πολιτών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άποψή του σχετικά με το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Αν δούμε δύο θέματα Μία ερώτηση ήταν ε, ότι ζητούσε από τους πολίτες να ε, θέσουν προτεραιότητες στο πώς μπορούμε να βγούμε από την, ε, από την κρίση. Το 29% είπαν να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες και τα δύο τρίτα των πολιτών είπαν ότι πρώτα θα πρέπει να τονώσουμε την οικονομία ή τουλάχιστον να το συνδυάσουμε και αυτό. Και όσον αφορά τις προτεραιότητες για τις πολιτικές, πάνω από το 50% των πολιτών και της Ευρώπης και της Ιρλανδίας είπαν ότι θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχουν λοιπόν, ε, υπάρχει διαφορά ε, απόψεων μεταξύ των ε, όσων λέγονται για την οικονομική κρίση και νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο κύριος Μπάτεν, ευχαριστώ πρόεδρε. Αύριο 23 Νοεμβρίου είναι η τέταρτη επέτειος του θανάτου του κυρίου Λιτβινέγκο στο Λονδίνο από πράκτορες του κρατικού του ρωσικού κράτους στα πλαίσια κρατικής τρομοκρατίας. Οι τρεις ύποπτοι, ο κύριος Λουγκαβόη, ο κύριος Κουρτσόν και ο κύριος Σοκολέγκο, είναι ακόμα ελεύθεροι στη Ρωσία. Ενώ η χείρα του κυρίου Λιτβινέγκο δεν μπορεί να ζητήσει την δικαιοσύνη. Δεν έχει γίνει ακόμα ανάκριση για την δικαστική έρευνα για την, το θάνατο αυτό. Ε, ζητώ λοιπόν από τις Βετανικές Αρχές να συγκαλέσουν άμεσα την ε, ανακριτική αρχή για να τεθούν φανερά οι αιτίες του θανάτου και να εντοπιστούν οι, οι υπεύθυνοι και να ζητηθεί από την αστυνομία να αναζητήσει τους δράστες. Ο κ. Λιτβινέγκο σκοτώθηκε σε βρετανικό έδαφος και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι το λιγότερο που μπορεί να διεκδικήσει η χείρα του. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμπόρσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πριν μία εβδομάδα η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της για την ενταξιακή διαδικασία των χωρών των Βαλκανίων. Δεν είναι σωστό να θέτουμε όρους για το ξεκίνημα των διαδικασιών και όταν τηρηθούν οι όροι αυτοί να μην ξεκινούμε ε, τις διαπραγματεύσεις. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε δίκαια τη Μακεδονία. Η Μακεδονία έχει πετύχει πολλά. 80% των νέων πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά από τα έξι τους. Η έκθεση της ε, Επιτροπής αναφέρεται στην πρόοδο ε, που έχει πετύχει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην σταθερότητα της διακυβέρνησης, στο σωστό πολιτικό διάλογο. Η Μακεδονία τήρησε όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αξίζει να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει να γίνει της διαδικασίας ένταξης στην Ένωση. Αλλιώς η Ένωση θα χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και όλων των άλλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρέιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην ε, χρηματοδοτήσει ε, ε, το, μεγάλο, μέσο διάσωση στη μάχη. Καταγγείλουμε τους, Βρετανούς, γιατί επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια στο θαλάσσιο του τομέα που βεβαίω είναι αυτός ο πιο πολύ στην περιοχή, θαλάσσια περιοχή του κόσμου. Οι εμπειρογνώμονε θεωρούν ότι η πρωτοποθέτηση σκαφών διάσωσης ε, θα επιτρέψουν την πρόληψη σοβαρών ε, ατυχημάτων. Αυτό θα διατηρήσει και το προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως πρέπει να χρηματοδοτείται από το κράτος να μην, να μην ιδιωτικοποιηθεί Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα και να ασχοληθεί η μεγάλη, με τη μεγάλη ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική την οποία διακηρύσει. Ο κύριος Ούτζας. Θέλω να ενημερώσω, ο κύριος Αούτζια, συγγνώμη, να ενημερώσω του ε, συναδέλφου ότι υποβάλαμε την ε, υπαριθμό 86 δημόσια δήλωση τότε στην προστασία του νερού ω δημόσιο αγαθού. Είναι ένα οικουμενικό αγαθό το νερό και η διαχείριση τη υπηρεσία ε, ε είναι πράξη ορθή διακυβέρνηση. Αυτή είναι οι, αυτές είναι οι βασικές αρχές, αρχές που κινητοποίησαν χιλιάδες Ιταλούς πολίτες να υποζητήσουν το δημοψήφισμα για την ε, αποφυγή της ιδιωτικοποίησης του νερού. Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι κομματική, αλλά είναι μια μάχη όλων. Η επιβεβαίωση κάτι τούτου θα γίνει, γίνεται από το γεγονός ότι συνάδελφοι διαφόρων πολιτικών ομάδων, πράσινοι, χρυσοσιαλιστές, ε, αριστερούς και ε, έχει τύχει μεγάλη υποστήριξη όλο το Κοινοβούλιο. Στόχος είναι να έχουμε πάνω από τις μισές υπογραφές μελών του Κοινοβουλίου για να γίνει επίσημη θέση του Κοινοβουλίου και να μπορέσει να προστατεύσει το νερό ως δικαίωμα και όχι ως κέρδος. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη. Οι πρόορες ε, κοινοβουλευτικές εκλογές ε, στη Μολδαβία θα αποφασίσουν για τις δημοκρατικές δυνάμεις στον κομμουνισμό. Οι δημοκρατικές δυνάμεις ε, είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ένταξης και τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί πρόοδοι οι οποίοι θα συνεχιστούν με αυτή την κατεύθυνση. Οι δημοκρατικέ δυνάμει θα πρέπει να παραμείνουν ενωμένε πριν και μετά τι εκλογέ. Οι εκλογέ τη Κυριακή θα πρέπει να είναι ελεύθερε ε, και ορθέ και οι εκλογέ πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Η βία του Απριλίου του 2009 δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η δημοκρατική κυβέρνηση δεν φτάνει στην εξουσία με τρομοκρατία και με εκλογική νοθεία θα ψηφίσει ο λαό τη μολδαβία την Κυριακή στι εκλογέ και όχι εμεί, αλλά εμεί υποστηρίζουμε το δημοκρατικό λαό εκφράζοντα αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκράντε Πασκουάλη έχει το λόγο. Πρόσφατα επιτέθηκαν και σκότωσαν 58 άτομα στην εκκλησία της Παναγίας στη Βαγδίτη. Μόνο και μόνο γιατί ήταν ε, στη Βαγδάτη, μόνο και μόνο γιατί ήταν χριστιανοί. Αυτό δεν είναι ένα απομονωμένο, μεμονωμένο γεγονός, αλλά το αποκορύφωμα επιθέσεων σε χριστιανούς στις ε, μουσουλμανικές χώρες, στο Μαρόκο, στην Τουρκία, στη Λιβύη, στην Αλγερία. Τον Ιανουάριο έξι χριστιανοί σφάχτηκαν στην πόρτα μιας εκκλησία στο Κάιρο. Μέχρι πότε θα παραμείνουν σιωπηλέ οι δυτικέ δημοκρατίες. Έκανε βέβαια ευτυχώ μια δήλωση ο κύριος Μπούσεκ, ενώ η καταδίκη τη κύρια Άστον ήταν καταδίκη τρομοκρατική επίθεση. Γιατί δεν αναφερόμαστε στο κίνητρο, το ότι ήταν χριστιανοί. Ο κύριο Καπατέρο δεν άκουσε τίποτα. Ο κύριο Ερντο, Ερντογάν δεν άκουσαν τίποτα. Τι η συμμαχία για τους πολιτισμούς, τι νόημα έχει. Τα ήξερε αυτά και τα έλεγε η Φαλάτσι όταν έλεγε ότι θα έρχουν οι Άραβες και κοντέψαν να τη λιθοβολήσουν. Θεός χωρέστην. Ευχαριστώ πρόεδρε. Grazie, la parola all'onorevole Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εκπαίδευση είναι μια προτεραιότητα στη στρατηγική για το 2020 και είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Αλλά η βουλγαρική κυβέρνηση ασκεί μια αντεθνική και αντιευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Η Βουλγαρία δαπανά μόνο 0,6% του ΑΕΠ της για την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη η Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών θα διαλυθεί και πρόκειται για ένα θεσμό που δημιουργήθηκε επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, επί Οθωμανικής κατοχής και από την Ακαδημία αυτή προέρχονται πολλοί επιστήμονες στη Βουλγαρία και αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βουλγαρική κυβέρνηση δεν βρίσκει δρόμο εξόδου από την κρίση, αντιθέτως επιλέγει την καταστροφή της παιδείας και του πολιτισμού. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι δεν κάνει ε, επαρκές, ε, επαρκείς διαβουλεύσεις οργανώθηκε την περασμένη εβδομάδα μία ακρόαση και φάνηκε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ε, για την καινούργια πρόταση οδηγίας και η Επιτροπή αρνείται να οργανώσει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ποια είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 40% των ε, ε, έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έργα χωρίς να αναφέρεται ο δημιουργός. Ε, είναι έργα ορφανά και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να διοργανωθούν οι σωστές διαβουλεύσεις. Ο κύριος Γκρότε. Οι δημοκρατικές η δημοκρατική διακυβέρνηση είναι ο πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι ε, επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι δημοκρατικές ε, και ε, ζητούν από συγκεκριμένη εταιρεία συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της μεταλλοβιομηχανίας. Αρνούνται όμως οι επιχειρήσει την παραχώρηση συμβάσεων εργασίας και κάνω έκκληση ε, προς την ε, επιχείρηση και προς τον επιχειρηματία τον κύριο Φιλιππόφ ε, να επανέλθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Με δημοκρατική συνεργασία θα πρέπει να καταλήξουμε σε καλύτερο και πιο δίκαιο σύστημα αντί να έχουμε κοινωνική δυσαρέσκεια και φόβο. Ένα τέτοιο σύστημα βλάπτει τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρέντε, ο κύριος Πρέντε έχει το λόγο. Δύο λόγια για τις ε, προεδρικές εκλογές στην ακτή Ελεφαντοστού, γιατί είμαι επικεφαλής της Επιτροπής Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Από τις αρχές Οκτωβρίου έχουμε στείλει 100 περίπου παρατηρητές από 26 χώρες, ολόκληρη την επικράτεια της ακτής Ελεφαντοστού. Η πρώτη σειρά, ε, ο πρώτος γύρος έγινε στις 31 Οκτωβρίου, σχετικά καλά, δεν υπήρχε απάτη βία. Ε, υπήρχε κάποια καθυστερημένη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εν γέννη όμως δεν υπήρξαν σοβαρά επεισόδια. Δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή και τα πράγματα έχουν, ε, ε, τα πνεύματα έχουν γίνει πιο ε, έντονα ε, υπάρχουν επιθέσεις ακόμα και εναντίον των παρατηρητών τους οποίους πολύ συχνά εμποδίζουν να κάνουν τη δουλειά τους και να παρακολουθήσουν την προετοιμασία της εκστρατείας. Πρέπει λοιπόν να ξαναεπικρατήσει ηρεμία ώστε να μπορέσει οι εκλογές να γίνουν κανονικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δε να προστατευθούν μέχρι την Κυριακή αλλά και μετά την Κυριακή παρατηρητές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στην έκθεση Μπέλετ, δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών ε, ε, εκπομπών για το μέλλον, το ψηφιακό μέλλον. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.